κοινοποίησαν πως ε, λόγω της κακοκαιρίας ε, της ε, προηγούμενης εβδομάδας υπλήξαν πάρα πολλοί πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είχαμε πλημμύρες, σφοδρές γενοπτώσεις και νομίζω πως όπως αυτό ζήτησαν και οι ομάδες θα συζητήσουμε αυτό το θέμα στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να εκφράσω εξ ονόματος σώματος την αλληλεγγύη μας στους πληγέντες και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να βοηθήσει γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία. 22 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε την δεύτερη διάσκεψη για το μέλλον της Συρίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. όπου θα έχουμε τους εκπροσώπους ε, του Συριακού Καθεστώτος και της Συριακής Αντιπολίτευσης με τους διεθνούς εταίρους με στόχο να βρεθεί ένας τρόπος να τελειώσει ο εμφύλιος και να σχηματιστεί μια μεταβατική κυβέρνηση. Η δύσκολη κατάσταση στην ε, Συρία βεβαίως δυσκολεύει τη διεξαγωγή της διάσκεψης αυτής, η οποία όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από όλους τους συμμετέχοντες να μην αναβάλουν την διάσκεψη, αλλά να παραβρεθούν. Τα... Οι κοινοβουλευτικές ομάδες ενέκριναν επίσης το αίτημα αυτό ομοφόνος και βέβαια θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε προσοχή τις εξελίξεις στην Συρία μέχρι να σταματήσει η σύγκρουση. Κυρίες και κύριοι, με πληροφόρησαν πως ο συνάδελφος Μπροκ δέχθηκε επίθεση από τον, λεκτική επίθεση από τον ε, Πρωθυπουργό της ε, Ρουμανίας για κάποιες δηλώσεις του που έκανε σχετικά με την μετανάστευση ε, εντός της Ένωσης και τον παρομοίασαν με Ναζί. Ανεξαρτήτως ε, του περιεχόμενου των δηλώσεων του κυρίου Μπρόκ, θεωρώ πως είναι απαράδεκτο πρώτο να γίνονται τέτοιες συγκρίσεις και βεβαίως δεύτερον νομίζω πως δεν τίθεται ζήτημα για την ακαιρεότητα του κυρίου Μπρόκ. Περνάω τώρα στις ανακοινώσεις. Το πρόγραμμα, το σχέδιο χρονοδιαγράμματος του 2015 είναι στην διάθεσή σας. Εγκρίθηκε η πρόταση αυτή από την διάσκεψη των Προέδρων. Τρίτη 14 Ιανουαρίου είναι η προθεσμία για τροπολογίες και Τετάρτη έχουμε την ψηφοφορία από τις αρμόδιες αρχές της Δανίας ε, πληροφορηθήκαμε πως εξελέγει ο κύριος Κλάους Λάρσεν Γένσεν, ο οποίος αντικαθιστά τον κύριο Γιώργενσεν με ισχύ από τις 13 Δεκεμβρίου 2013. Ο κύριος Γιώργενσεν έγινε υπουργό. Οι αρμόδιες αρχές Πολωνίας με ενημέρωσαν για την ε, εκλογή δύο συναδέλφων. Ο κύριος Μπιγνιέφ Ζαλέσκη, ο οποίος αντικαθιστά την κυρία Κολάρσκα Κολάρσκα-Μπομπίνσκα, και ο κύριος ε, Ταντέος Ρόστοιτ, ο οποίος αντικαθιστά τον κύριο Ραφάλ Τσασκόφσκι. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το άρθρο 4 επίσης ε, του κανονισμού οι συνάδελφοι αυτοί καταλαμβάνουν τους τους από τις 13 Δεκεμβρίου 2013 και βεβαίως ε, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 θα συμμετέχουν ε, με όλα τα δικαιώματα στη λειτουργία του Κοινοβουλίου μέχρι να εξεταστούν τα διαπιστευτήριά τους ε, και υπό την προϋπόθεση πως έχουν δηλώσει πως δεν υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο με τα καθήκοντα του Ευρωβουλευτή. Ο κύριος Godfrey Bloom φεύγει από την ομάδα EFD με ισχύ από 9 Ιανουαρίου 2014 και ανήκει στους μη εγγεγραμμένους. Το ΕΛΚ, οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Πράσινοι μου ζήτησαν ε, να ε, διορίσουν άτομα και να αλλάξει σύνθεση κάποιων επιτροπών και αντιπροσωπιών. Η λίστα είναι στην διάθεσή σας. Εάν μέχρι το τέλος συνεδρίας δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, εγκρίνονται αυτές οι αλλαγές.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 Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου συνυπέγραψα 18 νομοθήματα τα οποία εγκρίθηκαν με την τακτική νομοθετική διαδικασία. Όλα αυτά θα δημοσιευτούν στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης. Περνάμε τώρα στις εργασίες αυτής της ε, συνόδου. Κανείς δεν έχει προτείνει κάποια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ, κύριε Χουντή, για την ημερήσια διάταξη. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω κάτι στην ημερήσια διάταξη, αλλά επειδή είμαστε στο κομμάτι εκεί των ανακοινώσεων, θέλω να σας πω ότι κατά την τελετή έναρξης της ελληνικής προεδρίας... Äh, Μία στιγμή, κύριε Χούντι, να τελειώσουμε την ημερήσια διάταξη.